στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τώρα περνάω στις αλλαγές της ημερησία διάταξης. Η τελική ημερήσια διάταξη προσωρινή που υιοθετήθηκε στις 10 Νοεμβρίου βάσει του κανόνα 137 έχει διανεμηθεί και την έχετε όλη αυτή την προσωρινή ημερήσια διάταξη σχετικά την Δευτέρα και την Τρίτη δεν υπάρχει κανένα αίτημα για αλλαγή. Όσον αφορά στην Τετάρτη τώρα, σύμφωνα με όλες, ε, σε συμφωνία με όλες τις πολιτικές ομάδες, με την πλήρη συμφωνία όλων των πολιτικών μονάδων έχουμε τις ακόλουθες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος. Θα αρχίσουμε με δήλωση σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Το δεύτερο θέμα θα είναι προφορικές ερωτήσεις για το ανοιχτό διαδίκτυο. Το τρίτο προφορική ερώτηση για τους Ρωμά. Τέσσερα ε, δήλωση για την απαγόρευση πυρομαχικών διασποράς. Και πέμπτο θέμα προφορική ερώτηση για την νομοθεσία σχετικά με τον ΦΠΑ και την ψηφιακή αγορά τα άλλα θέματα στην, ε, στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης, στο, στο πρωί της Τετάρτης παραμένουν ως έχουν. Και θα ήθελα απλώ να επισημάνω ότι αυτές οι αλλαγές έγιναν σε συμφωνία με όλες τις πολιτικές ομάδες. Την Πέμπτη έχουμε δύο αλλαγές. Η πρώτη και πάλι σε συμφωνία με όλες τις πολιτικές ομάδες η δήλωση της Επιτροπής για την συμβολή της κοινή αλλιευτικής πολιτικής στην παραγωγή δημοσίων αγαθών αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη. Δεν θα υπάρξει δήλωση της Επιτροπής και επίσης την Πέμπτη και πάλι σε συμφωνία με όλες τις πολιτικές ομάδες σε σχέση με την εισήγηση του κυρίου Φλέκενστάιν για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, για την οποία είχε ε, προγραμματιστεί ψηφοφορία την Πέμπτη, οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν ότι δεν θα έπρεπε να γίνει ψηφοφορία για αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια αυτής της Συνόδου, αλλά να αναβληθεί η ψηφοφορία για τις 30 ε, Νοεμβρίου ή την 1η Δεκεμβρίου. Υπάρχει λοιπόν μια καθυστέρηση, μια αναβολή δύο εβδομάδων για αυτήν την ψηφοφορία και αυτό και πάλι η αλλαγή αυτή συμφωνήθηκε από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Αυτή αυτό είναι το πρόγραμμά μας για αυτήν την Ολομέλεια και μπορούμε να περάσουμε στο... Υπάρχει... Ο κύριος Πάσσαλτ ζητάει το λόγο. Ναι, πρόεδρε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα καλά, γιατί ακούσαμε μία φορά ότι η έκθεση Φλέκενστάιν θα αναβληθεί για τη μήνυ νομέλεια σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία και ε, μετά άκουσα ότι θα αναβληθεί και η συζήτηση. Παρακαλώ διευκρινίστε. Η ψηφοφορία, απαντάει ο Πρόεδρος, θα αναβληθεί. Δεν θα λάβει χώρα στην ολομέλεια αυτή, αλλά στην ε, επόμενη συνεδρίαση, 30 11 με 1η Δεκάτου. Εκεί θα γίνει η ψηφοφορία. Μάλιστα και έτσι ολοκληρώνονται λοιπόν ε, ε, τα θέματα περί ημερήσια διάταξης και περνάμε στο πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξη, ε, την έκθεση τη κυρία Αρακιάνη. Α, μπλε κάρτα, ζητάτε το λόγο. Ναι, να σας επιστήσω την προσοχή στο εξή. Θα ήθελα να πω ότι έχουν περάσει πέντε χρόνια μόλις από τότε που τα Ιρλανδικά αναγνωρίστηκαν στην Ευρώπη ως επίσημη γλώσσα και υπάρχει στο σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 22, 23 γλώσσες αλλά όχι στα Ιρλανδικά. Σας ζητώ να με βοηθήσετε. Πότε θα συμβαδίσει το Κοινοβούλιο με τα άλλα θεσμικά όργανα και θα φροντίσει να υπάρχουν επίσημες μεταφράσεις και στις 23 επίσημες γλώσσες. Για να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση καμίας γλώσσας. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπόδειξη αυτή. Θα εξετάσω το ζήτημα αυτό και θα σας αναφέρω τις εντυπώσεις μου. Σας ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να πω δύο λόγια, αν δεν έχετε αντίρρηση, και να υποστηρίξω αυτό που ανέφερε μόλις ο κ. Κάλλερ. Είναι πραγματικά ατυχές να αφήνετε κατά μέρο μία γλώσσα και θα ήθελα να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει και Πρόεδρος. Bo dzisiaj nie jestem w stanie Απάντησα ήδη στο αίτημα του κυρίου Γκάλερ ότι σήμερα στην παρούσα φάση δεν μπορώ να τοποθετηθώ, αλλά θα το εξετάσω. Διαδικαστικό, κύριε Ντεμπρούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επί του ιδίου θέματος. Όταν μιλώ εδώ στο Κοινοβούλιο, πάντα μιλώ, στη γλώσσα μου, τα ελληνικά. και οι ομιλίες μου είναι γραμμένες στα Ιρλανδικά. Τα κείμενα μένουν στα Ιρλανδικά μέχρι ότου μεταφραστούν στις άλλες 22 γλώσσες. Στην παρούσα, στη φάση μάλλον αυτή, εξαφανίζεται το αρχικό Ιρλανδικό κείμενο. Άρα το Ιρλανδικό κείμενο, το αρχικό, το πρωτότυπο κείμενο εξαφανίζεται από την ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και δεν μπορεί κανείς να το βρει. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, δεν μπορώ να πω όμω οτιδήποτε άλλο εκτό από αυτά που απάντησα στον κύριο Γκάλαγκερ. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Θα το εξετάσω προσωπικά. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρω ότι το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό και το αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα. Θα το εξετάσω. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έκθεση Σερακιάνη. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την εισηγήτρια να λάβει το λόγο. Η κυρία Σερακιάνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν σας εκθέσω τα περί της έκθεσής μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις που με βοήθησαν στην αναδιατύπωση του Σκούν Τρεμόσα ζήλ.